Uh, Συναδελφοί, καθίστε παρακαλώ, γιατί έχουμε αρκετή ψηφοφορία. Um, Συνάδελφοι, έτοιμοι. Έχουμε την ετήσια έκθεση σχετική με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Ο εισηγητή δεν επιθυμεί το λόγο, επομένω περνάμε απευθεία στην ψηφοφορία και ξεκινούμε με τη συμβαστική πρόταση 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14, άρχεται η ψηφοφορία τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16. Άρχεται. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 12. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 300, τροπολογία 362. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συνάδελφοι, προσοχή παρακαλώ. Συμβαστική τροπολογία 21, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 398, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της πληροφορίας. Εκρίνεται. 402. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 404. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 437. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 438. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 461, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 31, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 475, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 18, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 496. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε πληροφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 506. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 508. Μόνο για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 36, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 523, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία, Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 17, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 525. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 527. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 529. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 547. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 548. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 557, ε, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 568 και 578 είναι ταυτόσιμες. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Τροπολογία 575. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 581. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 582. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 583. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 593, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 596, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 20, αιτιολογικές εκθέσεις, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 38, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 24, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 23, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 25, άρχεται η ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορία. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 26, άρχεται η ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορία. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 28, άρχεται η ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Συμβαστική, εγκρίνεται, συμβαστική τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψυχοφορίας, Εγκρίνεται. Τροπολογία 187 και τροπολογία 188 ταυτόσιμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 35, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρυσι ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της Εγκρίνεται 41 ψήφοι υπέρ, 8 κατά και 3 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Έγγελ. Thank you, Mr. Engel. So now, colleagues, we move to the... Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στην απαλλαγή 2016. Κάτι έλεγα για καφέ, δεν έπρεπε να το έχω πει στο μικρόφωνο, λέει ο Πρόεδρος, αλλά αφού το είπα. Έκθεση. Σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικά του 2016. Ο κύριος Χρυσόγονος. Γενουσίγητης, θέλετε το λόγο ή να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Μπορούμε να ψηφίσουμε αμέσω. Λέω κύριο Χρυσόγονο. Ωραία, τροπολογία 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική αριθμό 1. Ψηφίστε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 9. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 10. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 11. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστικά παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. Εγκρίνεται με 45 ψήφους υπέρ, 5 κατά και μια αποχή. Περνάμε το επόμενο πάλι του κύριου Χρυσόγονου, άλλη μια απαλλαγή, Οργανισμός Ευρωπαϊκή Ένωση για συνεργασία στο Μέτρη τη του νόμου, Europol. Ψηφίζουμε ένα, υπέρ, ε, ψηφίστε μάλλον, πέρας, εγκρίθηκε. Συμβαστική αριθμός ένα. ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 2, συμβαστική δύο. Ψηφίστε, πέρας, Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ψηφίστε. 9. Πέρας. Απορρίπτεται. 10. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. 15. Ψηφίστε παρακαλώ. Α, 15. Ή όχι. όχι, καταπίπτει 15. Οπότε πάμε απευθεία στη συμβαστική 4. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. 18 τώρα. Ψηφίστε. 18 που μιλάει για τις δράσεις της Γιουροπολέ. Τέλος, εγκρίθηκε. Τροπολογία 20. Χωρίς το τμήμα που λέει ότι λυπάται επειδή και τα λοιπά. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 20, το τμήμα που λέει ότι λυπάται που η δημοσίευση είναι σε κρεμότητα κτλ. Ψηφίστε. Η τροπολογία 20. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τελική ψηφοφορία ονομαστικά. Ψηφίστε. Πέρας. Και εγκρίθηκε 46 υπέρ, 5 κατά και μία αποχή. Περνάμε στην επόμενη απολογή Eurojust αυτή τη φορά, συμβαστική 1. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 2. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 7. Ψηφίστε. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συμβαστική αριθμός 3. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τώρα τελική ψηφοφορία ονομαστικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε 46 υπέρ, 6 κατά καμία αποχή. Περνάμε στην απαλλαγή της Frontex. Συμβιβαστική αριθμό 1. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία Τέσσερα. Το κομμάτι που λέει αναγνωρίζει τον προπολογισμό της υπηρεσία. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 3. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Το δείγμα που λέει σημειώνει επ' αυτού για το προσωπικό κλπ. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 13. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 4. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 5. Ψηφίστε. 5. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 6. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τελική ψηφοφορία ονομαστική τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τελική ψηφοφορία, ναι, για τη Frontex, έτσι. Ψηφίστε παρακαλώ. Τελική ψηφοφορία, τέλος. Εγκρίθηκε 42 υπέρ 7 κατά 3 αποχές. Το ΕΛΚ προσπαθεί να μου πει κάτι. Κλοντ, να μιλάς στο μικρόφωνο παρακαλώ, γιατί πολλές φορές κοιτάς τον κατάλογο σου και εμεί δεν σε ακούμε καλά. Και μερικά πράγματα είναι πολύ λεπτά, έτσι, του δευτερόλεπτου και κάτι λες, εγώ δεν το βλέπω, οπότε παρακαλώ να μιλάς στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο, αυτό μόνο ζητάω. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Θες να μιλώ πιο δυνατά πιο δυνατά. Καλά, θα μιλώ πιο δυνατά και θα απευθύνομαι στο μικρόφωνο. Βέβαια και εγώ ψηφίζω, όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει. Θα φροντίσω να μιλώ πιο δυνατά. Συγγνώμη. Μπορεί να μην σας αρέσει να μιλάω ακόμα πιο δυνατά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, επόμενη απαλλαγή τώρα που θα εξετάσουμε είναι Να, με μπερδεύσατε τώρα. Και δεν ξέρω που βρίσκομαι. Λοιπόν, συναδελφοί. Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροπολογία αριθμό 1. Ψηφίστε παρακαλώ, με πιο δυνατή φωνή τώρα. Στο μικρόφωνο μιλάω. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική αριθμός 1. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. 7. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική α, όχι, μια στιγμή διορθώνει ο πρόεδρος. Πρέπει να ψηφίσουμε τροπολογία 10 τώρα. Ψηφίστε. Τροπολογία 10, ναι. Βλέπετε, δεν θα το ξανακούσω γιατί δημιουργεί χάος εδώ πέρα. Έλεγα τροπολογία 10. Τελειώσαμε την ψηφοφορία και απορρίφθηκε. Καλά, θα επιστρέψω στην κανονική μου φωνή, γιατί άμα μιλάω πιο δυνατά μπερδευόμαστε. Λοιπόν, συμβαστική 5, ψηφίστε. Α, όχι, να, πάλι μπερδεύτηκα. Έχουμε τις τροπολογίες 8 και 9. Ψηφίστε παρακαλώ. Έχασα το ρυθμό μου. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Συμβαστική 5 τώρα. Έτσι. Συμβαστική 5. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τελική ψηφοφορία ονομαστικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Με 43 υπέρ, 7 κατά και μια αποχή. Τώρα, απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Τροπολογία αριθμός 1. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 2. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 3. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 4. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 5. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική αριθμό 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 2. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία τώρα, τελική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε 45 υπέρ, 5 κατά και μία αποχή. Και τώρα περνάμε στην απαλλαγή της ΣΥΠΟΛ. Τροπολογία αριθμός 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίφθηκε 2. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τρία. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Πέντε. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική αριθμός 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική αριθμός 3. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίνεται. 13. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Και εγκρίθηκε. 46 ψήφοι υπέρ, 5 κατά και μία αποχή. Επόμενη απαλλαγή τώρα είναι της ΕΑΣΟ. Και αρχίζουμε τη συμβαστική αριθμός 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 2. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 3. Άρχεται. Περάς. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Ε, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται. Συμβαστική 6, άρχιτε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 8. Είπε ε, ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Απαλλαγή 2016 για το EU Lisa, συμβαστική 1, αν είστε έτοιμοι όλοι, συμβαστική 1. Εγκρίνεται σημαντική 2. Άρχεται. Πέρας. Συμβαστική 3. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 8. Ψηφίστε. Τέλος. εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Όχι. Έκανα λάθος. Συμβαστική 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τώρα τροπολογία 11 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 12 ε, άρχεται. Για ένα λεπτό. Ε, πέρας για την 12. Απορρίπτεται 13. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 15. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 16. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 23. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 8. Έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 28. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 29. Έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 30. Έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ονομαστική. Έρχεται. εγκρίθηκε 45 προς 6 καμία αποχή απαλλαγή τώρα για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασία Δεδομένων Συμβαστική 1. Ενάρτητα. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 2. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. σημαντική 3 Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. σημαντική 4 Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 9 Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται 10 Πες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 6 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική με ονομαστική άρχεται. Πέρας. 46 προς 6, καμία αποχή εγκρίνεται. Γενικό Προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση, Απαλλαγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, σημαντική ένα. 1. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρα Απορρίπτεται. Συμβαστική 1, τμήμα 1, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1, τμήμα 2, άρχεται. Πέρασε Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ονομαστική άρχεται. 45 ψήφι προς 6, μία αποχή. Κύριε Χρυσόβουλο, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ε, γεια σας συνάδελφοι, ένα λεπτάκι. Διακόπτουμε για μισή ώρα και μετά και κλεισμένο των θυρών. Για όσους θέλουν και όσους δεν θέλουν, το Σαββατοκύριακο.